Γεια σας. Επανερχόμαστε στην ε, συνεδρίαση. Ως συνήθως έχουμε την παρουσίαση της μελέτης εφαρμογή του συστήματος αποκλήσεων από τους κανόνες προέλευσης για τα αλληλευτικά προϊόντα στην Παππούα Ζία, Νέα Γουινέα και τη νήσους Φίτζη. Χωρίς περαιτέρω εισαγωγή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΣΥΝΤΑ, τον κύριο Μορέιρα που είναι μαζί μα. Τον κάλεσα να έρθει σήμερα το απόγευμα εδώ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι εδώ, όπως και όλα τα άλλα μέλη της Επιτροπής Ίντα εδώ. Πρόκειται για μια καλή αρχή σε σχέση μεταξύ της Επιτροπής Ίντα και της Αλίας, που πολλές φορές έχουν περισσότερα κοινά σημεία από ό,τι φαίνεται αποφάσεις οι δράσεις της ΙΝΤΑ έχουν σημαντικές επιπτώσεις πολλές φορές στην Επιτροπή Αλίας. Γι' αυτό καλύτερα να έχουμε από κοινού σχέση και να προχωρούμε από κοινού παρά ο καθένας να ακολουθεί το δρόμο του και να γίνονται τα πράγματα πιο πολύπλοκα και να καταλήγουμε σε καταστάσεις μη επιθυμητές. Αν είχαμε καλύτερη επικοινωνία θα ήταν καλύτερα. Γι' αυτό θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΙΝΤΑ, τον κύριο Μορέιρα, και να πω ότι αισθάνεται η Επιτροπή μας ότι θα πρέπει να έχουμε πιο στενή σχέση, να έχουμε μια αγαστή συνεργασία και σχέση μεταξύ των δύο Επιτροπών και επαναλαμβάνω, αυτό είναι απαραίτητο δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία μέσω των, επιτρο... των ε, συμφωνιών που υπογράφει η ιτρί και έχουν ε, επιπτώσεις για μας. Αυτό είναι λοιπόν ένα σαφές παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Γι' αυτό εξ ονόματος όλης τη Επιτροπής θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Μορέιρα που είστε εδώ. Όντως πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Στην αρχή του έτους αναθέτηκε, ανατέθηκε εξωτερική μελέτη για την εφαρμογή του συστήματος αποκλήσεως. Ολοκληρώθηκε πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Ήδη έχει διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους αυτής της Επιτροπής και βεβαίω τη μελέτη είναι στη διάθεση όλων όσων θέλουν να τη μελετήσουν. Δίδω στο το λόγο στον κύριο Μορέιρα, αλλά θα θέλαμε να καλωσορίσουμε και τους συντάκτες αυτής της μελέτης, τον κύριο Αντώνιο Σάνθ, που θα κάνει την εισαγωγή στη μελέτη αυτή και μετά τους κυρίους Πίκοκ, Μπούς και την κυρία Μίλλερ από το Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας που θα μας παρουσιάσουν την μελέτη που έκαναν και μετά βεβαίως θα αρχίσει η συζήτηση και θα μπορούν να παρέμβουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι. Έχουμε περίπου μια ώρα στη διάθεσή μας, αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε ήρεμα να συζητήσουμε την ε, έκθεση αυτή τη μελέτη. Ο κύριος Σάντς, ο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Όπως σας είπα, θα παρουσιάσω αυτή την έκθεση σήμερα μαζί με κάποιους εμπειρογνώμονες, την Άγγελ Πίκα, ε, τον επικεφαλής της μελέτης και τον εκπρόσωπο του ε, Πανεπιστημίου, τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου που θα εξετάζουν τα ζητήματα διακυβέρνησης. Το περιεχόμενο αυτής της ε, παρουσίασης είναι μια παρουσίαση της μεθοδολογίας και παρουσίαση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων δεδομένου του μικρού χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας. Η παρουσίαση θα εστιαστεί στις οικονομικές επιπτώσεις και στα ζητήματα διακυβέρνησης ε, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μελέτης επιπτώσεων. Θέλαμε μέσω αυτής της μελέτης να παρουσιάσουμε μια ανεξάρτητη ανάλυση των επιπτώσεων στο πλαίσιο της οικονομικής ε, συμφωνίας, της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παπουάς Νέας Γουινέας, καθώς και τις περιβαλλοντικές ε, και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις στη βιομηχανία τόνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνεργάτε σε αυτή τη μελέτη ήταν Biomaker και Σάντ στο Κέντρο Θαλασσών Επιστημών στο Αλγκάρβε, το Πανεπιστήμιο του Βίγου και το Πανεπιστήμιο του Βάχενίγκεν στι κατοχώρε. Ε, διερκέσει η μελέτη έξι μήνες. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή αυτή τη μελέτη, βασίστηκε σε ε, ε, έρευνα και σε οικονομετρικές αναλύσεις, επίσης διαβουλεύσεις με ενδιαφερομένους. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν διαθέσιμες για συναντήσεις. Άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι η βιομηχανία με κυβερνητικοί οργανισμοί και διεθνείς οργανισμοί. Τέλος, στο πλαίσιο της μεθόδους μας, τρεις εμπειρογνώμονες ε, της ομάδας μας επισκεφτήκαν τη χώρα και εστιάστηκαν στι συναντήσεις με αρχές της Παππούας Νέας Γουινέας, διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ε, την Παγκοσμία Τράπεζα και με κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και ε, διάφορους τομείς της βιομηχανίας της χώρας. μερικά λόγια τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο της μελέτης. Τι αφορά αυτή η εξαίρεση, γνωστή ως Global Sourcing, επιρρεπεί τη χρήση πρώτων υλών που δεν προέρχονται από τη χώρα, αλλά που εκφορτώθηκαν σε ένα λιμένα της χώρας, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ινέα. Αυτές οι εξαιρέσεις ισχύουν από το Μάρτιο 2008 λόγω του γεγονότος ότι έχει πολύ τόνο αλλά όχι ε, ικανότητα στόλου. Δηλαδή μπορεί να υποφεληθεί η Παπουανέγουινη από τους σπόρους ε, εφόσον μόνο ε, γίνει η κατεργασία του τόνου στην ίδια τη χώρα. Η Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία, για τη βιομηχανία τόνου, καθώς και κοινωνικές επιπτώσεις ε, και επιπτώσεις για το περιβάλλον στην Παπουανέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξήγησε ότι αυτή είναι μια εξαιρετική ε, περίπτωση εξαίρεσης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις η βιομηχανία τόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την Επιτροπή Αλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζουν την απόκληση, αλλά ορισμένοι εξέφρασαν ανησυχίε όσον αφορά τι επιπτώσει για τον τόνο και κάποιοι άλλοι σε σχέση με τη συμμορφούς με τα εργασιακά δικαιώματα. Σε αυτές τις διαφάνειες σκοπός είναι να σας δώσουμε μερικά νούμερα, για να, μερικά ψωστά για να δείτε την ευρύτερη εικόνα τα λεύματα των αντιστοιχούν 10% ε, στην Παπούα σε σχέση με το σύνολο του Δυτικού Κεντρικού Ειρηνικού. Και από άποψη εμπορική, οι εισαγωγές ε, τόνου από την ε, Παπούα αντιστοιχούν σε 5% των συνολικών εισαγωγών. Τώρα δίνω στον Νάιτζελ τον λόγο για την οικονομικό σκέλος. Καλησπέρα, είμαι ο Νάιτζελ Πίκοκ και εγώ διεξήγαγα την οικονομική εκτίμηση επιπτώσεων για αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη. Δύο ερωτήματα κλειδιά τέθηκαν από οικονομική άποψη. Πώς αυτή η απόκληση οδήγησε σε οδήγηση της ε, ικανότητας ε, παρασκευής, της ικανότητας μεταποίησης στη χώρα, αυξάνοντας την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και το οικονομικό όφελος για την νέα, είναι το άλλο. Ερώτημα κλειδί είναι κατά πόσο υπήρξαν αμοιβαία ε, μειονεκτήματα για τις βιομηχανίες μεταποίησης τόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα, κατά πόσο λοιπόν αυξήθηκε η μεταποίηση στην παππούα Γουινέα μετά από την εφαρμογή της απόκλησης. Όχι ακόμα. Η παραγωγή είναι περίπου 30.000 τόνους ε, ε, που χρειάζεται περίπου 60.000 τόνους να εισέρχεται στις βιομηχανίες ε, μπορούν να μεταποιήσουν περίπου 500 τόνους την ημέρα οι βιομηχανίες αυτές. Αλλά πιστεύω το σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι η ανάπτυξη μιας μεγάλης βιομηχανίας χρειάζεται 10 με 20 χρόνια ε, σε ανεπτυγμένες χώρες όπως την Ευρώπη, σε ένα μέρος όπως την Παππούα, Νέα όπου οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, πιθανώς θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Συνεπώς είναι πρόημο το να προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τέτοιες επιπτώσεις. Ωστόσο, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι τα πράγματα αλλάζουν. Σε αυτή τη φωτογραφία, στη διαφανεία, βλέπετε ένα μεγάλο εργοστάσιο μεταπίσης που ε, χτίζεται στη Μαλαχάγκ, σε ε, μια αστική περιοχή της Νέας ε, Είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό εγχείρημα το να προσπαθήσουν να εγκαταστήσουν ένα εμπορικό κέντρο μια, ένα βιομηχανικό κέντρο μάλλον, μια μαλαισιανή εταιρεία, έχει χτίσει ένα εργοστάσιο μεταποίησης τόνου, η Dongwon από την Κόρεα, μία από τις μεγαλύτερες ε, αλληλευτικές επιχειρήσεις ε, του κόσμου και η Χαλισέγγα από την κινή. έχουν δεσμεύσει πολλές επενδύσεις ε, στη μεταποίηση τόνου εκεί και μετά στο Μαντάγκ άλλη παράκτια πόλη της Παπούας, ε, η, εκεί Νιουτζίνη Τούνα υποτίθεται ότι θα επενδύσει σε μια βιομηχανική ζώνη που επιχειρείται να αναπτυχθεί στην ε, ακτή. Όλες μαζί αυτές οι δεσμεύσεις ε, δείχνουν σημαντική αύξηση της παραγωγής τόνου, ε, σε κονσέρβα και, και καρέ τόνου. Η, η πρώτη ύλη που θεωρείται ότι θα αναπτυχθεί από 70 τόνους την ημέρα σε 360 καθώς ε, αυξάνουν τη χωρητικότητά τους στα υπάρχοντα ε, υπάρχουσες βιομηχανίες ε, και αυξάνουν το, την εισρωή πρώτων υλών. Έτσι θεωρείται ότι βάσει όλων αυτών των επενδύσεων του χρόνου θα είναι 90.000 τόνοι με αύξηση 600 τόνων ανά ημέρα. Βλέπετε το αποτέλεσμα στο παρακάτω γράφημα. Βλέπετε 90.000 τόνοι αναμένονται για του χρόνου έως 240.000 τόνους αύξηση το 2018. Δηλαδή αύξηση από 50.000% ε, τόνων προϊόν τόνου προϊόντος έω 124.000 τόνου προϊόντος. Ποια είναι τα ωφέλη για την Παπούα. Πρώτα απ' όλα επενδύσει που ήδη λαμβάνουν χώρα. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία γι' αυτό, απασχόληση, αναμένεται να αυξηθεί από 5.800 σήμερα σε 20.000 μέχρι το 2018 και ως επιτοπλίστων γυναίκες εισοδήματα συμβάλλει στην οικονομία από 21 εκατομμύρια σήμερα δολάρια σε, ε, αναμένεται να αυξηθεί σε 70 εκατομμύρια τώρα, οι δραστηριότητε ε, ε, έναρξης ε, πιστεύετε ότι θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας σε διάφορες περιοχές για την υποστήριξη των εργοστασίων μεταπίσης τόνου από 2.600 άτομα σε 5.000 άτομα μέσα στο 2020 Επίσης φόροι που θα ε, εισπράξει η κυβέρνηση πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικό. Θα αποτελέσει ένα κέντρο ε, ε, οικοδόμησης κρίσιμης οικονομικής μάζας, ειδικότερα στο ΛΑΕ και θα δημιουργήσει και άλλες βιομηχανίες υποστήριξης, μηχανική μηχανικής και υπηρεσιών ώστε να υποστηριχθεί αυτή η οικονομική δραστηριότητα σε, αυτή τη μηχανική ζώνη της Παππούας, Νέας Γουινέας. Για να μιλήσουμε τώρα για την αξία την αξία προτίμησης, ε, την προτιμησική αξία. Εδώ σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε το κόστος παραγωγής που έχουμε αναλύσει σε τρεις αγορές. Κοιτάξαμε την Παππού, Νέα την Ταϊλάνδη ως την πρώτη χαμηλού κόστους παραγωγική χώρα και στον Ισημερινό. Ο Ισημερινός επειδή αποτελεί σημαντικό προμηθευτή της ευρωπαϊκής αγοράς αυτό που είδαμε είναι ότι το κόστος, το αρχικό κόστος πρώτης ύλη είναι το ίδιο περίπου για όλες τις ε, χώρες, αλλά το κόστος μεταποίηση είναι πολύ μεγαλύτερο, σχεδόν διπλάσιο στην Παπουανέου είναι. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η προτιμησιακή πρόσβαση είναι κρίσιμη σημασία. Όταν βλέπει κανείς το κόστος ε, στην Ταϊλάνδη, ε, καταλήγουμε σε τελικό κόστος μαζί με το φορό 33 περίπου ευρώ το οποίο είναι περίπου ίδιο, ίσο με το κόστος της Παππούας Νέας Αλλά πραγματικά ε, αυτό δείχνει ότι απαιτείται να υπάρχει προτιμησιακή πρόσβαση για την Παππούα Νέα Από την άλλη πλευρά, η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμη σημασία για την Παππούα Νέα αν το χωρίσουμε στις τρεις κατηγορίες ε, προϊόντων, ε, κατεψυγμένο τόνο, φιλέτα τόνου, ή καρέ τόνου όπως λέγονται, και στο κάτω-κάτω βλέπετε τις κονσέρβες τόνου. Η μεγαλύτερη ποσότητα κατεψυγμένου τόνου πηγαίνει στις Φιλιππίνες, αλλά από τα φιλέτα, από το καρέ τόνου, τα περισσότερα πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως επιτοπλίστων στην Ισπανία, και γενικώ οι μπλε περιοχές που βλέπετε στα γραφήματα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και όπω βλέπετε ε, σχεδόν όλε όλες οι κονσέρβες των πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω στη Γερμανία. Η αγορά λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική για την Παπουανεγουενία με δύο τρόπου Πρώτα απ' όλα λόγω τη προτίμηση, διότι εκεί πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρο των προϊόντων, αλλά είναι μια σύμμετρη σχέση, επειδή η είναι, είναι πολύ λιγότερο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα δύο γραφήματα δείχνουν πρώτα την αγορά των καρετών, των φιλετών τόνου και εκεί βλέπετε ότι η Λατινική Αμερική είναι μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής φιλετών τόνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω-κάτω, εκεί που δείχνει το βέλος, βλέπετε μία γραμμή σε αύξουσα πορεία. Είναι η Παπώνε Γουινέα που είναι δεν είναι πολύ μεγάλος προμηθευτής. Στο δεύτερο γράφημα βλέπετε ο κονσερβοποιημένο τόνο και ο κύριος προμηθευτής αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή της ε, Αφρικής, ε, της Καραβικής και του Ειρηνικού. Ουσιαστικά μειώνεται η προμήθεια από αυτή την περιοχή. Ε, γίνεται σχεδόν... Μετά έχουμε την Ανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και κάτω-κάτω βλέπετε την Παπουανέα Γουινέα, που είναι μικρός παραγωγός αλλά σημαντικός. Η Παπονεγουίνα λοιπόν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντική η Ευρώπη για την Παππού, αλλά η Παπονεγουίνα είναι μικρό προμηθευτή για την Ευρώπη. Η Παπονεγουίνα υποφελείται εξαιρετικά από αυτό το εμπόριο. και είναι τα πιθανά μειονεκτήματα για τη βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει της οικονομικής ανάλυσης που έγινε στο πλαίσιο της μελέτης, εξετάζοντας ε, τάσεις ε, και στοιχεία και μελέτη συσχετισμού, αυτό που αναγνωρίστηκε σε ιστορική βάση είναι ότι θα υπάρξει κάποιο μειονέκτημα. Δύο σενάρια διαφαίνονται. Το πρώτο είναι το πιο ευνοϊκό, όπου αυξάνεται η ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παπουανέγου είναι αυξάνει κατά 10% τις εξαγωγές της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λιγότερο ευνοϊκό είναι αύξηση των εξαγωγών της Παππούας Νέας κατά 20% και η ζήτηση της Ευρώπης να μειώνεται. Στην πρώτη περίπτωση ε, μειώνεται κατά 1% η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δηλαδή με μη απώλεια αξία 5,2 εκατομμυρίων και απώλεια 180 θέσεων ε, Στο δεύτερο σενάριο που δοκιμάζεται και στο πλαίσιο της μελέτης βλέπουμε μείωση παραγωγής κατά 7% μείωση της προστιθέμενης αξίας κατά 43 εκατομμύρια και απώλεια 1.500 θέσεων εργασίας. Η μελέτη, αυτή η οικονομετρική μελέτη εξετάζει επίσης και τρίτες χώρες που είναι πολύ πιο δύσκολες για λόγω των ιστορικών εμπορικών δεδομένων και βλέπουμε μια ανάμεικτη εικόνα θετικών και αρνητικών συσχετισμών. Αυτό που είναι σημαντικό να δούμε είναι η γενικότερη βιομηχανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα φιλέτα τόνου. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα υψηλά εργατικά για την παραγωγή του κονσερβοποιημένου τόνου έχει εκχωρηθεί σε χώρε χαμηλότερου εργατικού κόστου. Έτσι, οι ευρωπαϊκέ βιομηχανικέ διαδικασίε ε, συνεχίζουν με επιτυχία. Αυτό που βλέπετε στο πάνω γράφημα είναι τη μείωση του... των εισαγωγών ε, ομού ολόκληρου τόνου που πέφτει τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, η πορτοκαλή πλευρά που είναι τα φιλέτα ευξάνεται και φαίνεται να υπάρχει κάποιο συσχετισμό μεταξύ αυτών των δύο. Πιο κάτω βλέπετε μια πιο ασθενή γραμμή που δείχνει την κατάσταση στην Ισπανία που είναι η πιο σημαντική χώρα μεταποίηση τόνου στην Ευρώπη και που ακολουθεί την ίδια πορεία με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι στο πανό γράφημα βλέπετε ουσιαστικά ολόκληρους, αφορά ολόκληρους τόνους ε, και τα φιλέτα τόνων. Αυτή η σύγκριση γίνεται. Ε, στο κάτω γράφημα βλέπουμε τον τρόπο που αυξάνεται η ζήτηση για φιλέτα, για καρετόνου και όπως βλέπετε θα επαναμένεται σημαντική αύξηση της ζήτησης. Ε. Η Ισπανία ειδικότερα συμβάλλει σε αυτή την ε, αύξηση των εισαγωγών ε, καρετών. Έτσι λοιπόν η Παπώνα γίνεται σημαντικός προμηθευτής ε, σε αυτό το γράφημα. Βλέπετε τις εξαγωγές τόνου από την Παπούα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλες επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση. Ο κονσερβοποιημένος τόνος έχει αυξηθεί και έχει φτάσει σε μια η ισορροπία είναι η πάνω καμπύλη. Ο κατεψυγμένος δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα, αλλά αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η καμπύλη των φυλατών τόνου, των τόνου, που έχουν σημειώσει πολύ πρόσφατα πολύ μεγάλη αύξηση. 80% πηγαίνει στην Ιταλία, 19% πηγαίνει στην Ιταλία. Και η Παπώνα Γουενέχη έχει γίνει σημαντικός προμηθευτής καρετόνου ενώ ο κονσερβοποιημένο τόνος είναι ανταγωνιστή για τι μεταπητικές βιομηχανίες στην Ευρώπη ενώ τα φιλέτα τόνου είναι αυτά που επιτρέπουν στι ευρωπαϊκές βιομηχανίες να συνεχίσουν τι δραστηριότητε του. Ε, ένα ζήτημα είναι τα ζητήματα υγιεινή, τα SPS ε, όπω αναφέρονται. Αυτό ξεκίνησε το 2008, όπου ο κονσερβοποιημένο τόνος απαγορεύτηκε να απολύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιο διάστημα. Το SPS λοιπόν έχει τεθεί ο ζήτημα σε αυτή τη μελέτη και το εξετάζουμε στο πλαίσιο της μελέτης και τότε γρήγορα τις γρήγορες συναγερμούς, τους ταχύς συναγερμούς. Τις έγκαιρες προειδοποιήσεις. Και βλέπουμε ότι για κάποια στιγμή νομίζω ότι τα πράγματα πήγαιναν χειρότερα. Αλλά όπως βλέπουμε στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα ήταν σε κατεψυγμένο τόνο, φιλέτα ή κατεψυγμένο τόνο που είχε αποσταλεί σε αυτές τις ε, συνθήκες σε κοντέινερ ψυγεία για την Ευρώπη. Αλλά το, το πρόβλημα δεν ήταν κάτι που υπήρχε στα μεταποιητικές βιομηχανίες στην Παπουανέου αλλά είχε παρουσιαστεί κατά τη μεταφορά. Αυτό δεν σημαίνει Τώρα, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου. thanks very much, Nigel. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λέγαμε Σάλαμ Μπούς Είμαι καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο και είχαμε ορισμένα input όσον αφορά αυτή τη ε, μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση της αλίας του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού σε σχέση με το CPC. Ο στόχος της παρουσίας, και θα είμαι αρκετά σύντομος γιατί έχουμε ξεπεράσει την ώρα μας, είναι να δείξουμε το σύνθετο περιφερειακό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει η χώρα η διαχείριση του τόνου στο Δυτικό Ειρηνικό και να προσπαθήσουμε να εξολογήσουμε τη σχέση αυτή ε, μεταξύ WCPFC και PA. Ε, έχουμε λίγα μέλη τα οποία έχουν διάφορα δικαιώματα και ευθύνες για να παρέχουν κάποιες, ε, να δίνουν κάποιες ιδέες στη διαδικασία λήψης απόφασης. Η Παπούα Νέα Γουινέ έχει σημαντικό ρόλο. Ε, βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια και είναι το 80% των ελευμάτων σε αυτή την περιοχή και 8,5% των συνολικών αλλιευμάτων προέρχεται από τον εθνικό στόλο στην, ε, της Παππούας Νέας Γουινέα. Ο, κεντρικό κεντρικός και δυτικός ειρηνικός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και αυτό το ευρύτερο πλαίσιο απαρτίζεται από τις διάφορες ε, συνθήκες που οδηγούν στη συλλογική διαχείριση και επίσης οι, οι συνθήκες αυτές χρησιμοποιούνται ώστε να ανεχθεί κάποιος έλεγχος ε, στα, στην αλία. Και υπάρχουν διάφορες άλλες ε, ομάδες, τα PNA, και υπάρχουν άλλες υποπεριφερικές ομάδες ε, οι οποίες ε, αφορούν τις διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά την αλία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την περιοχή αυτή χωρίς να μιλήσουμε για τη σύνθετη λεπίδραση μεταξύ των χωρών μελών και μεταξύ των ε, πιο απομακρυσμένων ε, χωρών που αλλιεύουν σε αυτά τα ύδατα. Όσον αφορά τα αποθέματα του τόνου, μπορούμε να κεντρωθούμε σε τρία είδη και την σχέση μεταξύ τους. Ο κεντρικός και δυτικός ειρηνικός ε, φτάνει στα όρια της βιώσιμης εκμετάλλευσης, αλλά αυτό αφορά μόνο ορισμένα είδη. Η παραγωγή παραμένει εντός βιώσιμων ορίων. Ε, και έχουμε εδώ το μονόφαλμο τόνο ε, και τον κυτρινόπτερο τόνο, που δεν έχει φτάσει σε επίπεδα υπεραλίευσης. Η παλαμίδα είναι μεταξύ 70 και 85% του συνόλου των ελευμάτων και παραμένει λοιπόν εντός των βιώσιμων ορίων. Ο στόχος του WCPFC όσον αφορά τη συντήρηση είναι να μειωθεί η θνησιμότητα του μεγαλόφθαλμου και του κυτρινοπτερού τόνου κατά 30%. Δηλαδή κατά το του 2004. Μία αναθεώρηση του WCPFC έγινε ε, μεταξύ του 2010 και το 2011 και έγινε μία αξιολόγηση και ε, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα του WCPFC. Το άρθρο 6 εξετάζει πόσο αποτελεσματική ήταν η WCPFC όσον αφορά την κατάρτιση σημείων αναφοράς, όσον αφορά την εφαρμογή κάποιων αρχών πρόληψης, που είναι μια βασική, ένας βασικός στόχος της πολιτικής. Δεύτερον, ήταν να εξεταστούν οι διάφορες διαπραγματεύσεις που γίνονται όσον αφορά τις εξαιρέσεις από διάφορες περιοχές και από το επίπεδο της εθνικής δικαιοδοσίας. Και γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τα διάφορα μέτρα διαχείρισης του πλήρους φάσματος των αποθεμάτων. Και υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των χωρών του ειρηνικού ε, και άλλων ε, χωρών. Τώρα, οι εξαιρέσει που περιλαμβάνουν την Παππούα Νέα Γουινέα θεωρούνται ω βασικό πρόβλημα τη διαχείριση των αποθεμάτων όσον αφορά το πλήρε φάσμα του και αυτέ οι εξαιρέσει περιλαμβάνουν συνεχή πρόσβαση για στόλου ε, σε χώρε του ειρηνικού. Ε, δεν υπάρχουν ε, ε, όρια όσον αφορά την αλίευση του, μονόφθαλμου, του μεγαλόφθαλμου τόνου με τα παραγαδιάρικα Ε, και ε, υπάρχουν, υπάρχει εφαρμογή του Vessel Day Scheme για ορισμένε χώρες ε, και αφορά τα σκάφη των εν χωρών. Τέλος, υπάρχει ένα άλλο θέμα που αφορά τον επιμερισμό των ημερών, αλλιώς όσον αφορά αυτό το ε, σχήμα, το Vessel Day Scheme, ε, και τον αριθμό των ημερών που έχουν επιμεριστεί στα διάφορα λευτικά σκάφη και έχει εξελιχθεί το σύστημα αυτό αποτελεσματικό και έχουν ε, γίνει και κάποιες βελτιώσεις. Ένα περαιτέρω θέμα αφορά το IUU και αυτό ε, έγινε αντικείμενο διαφόρων αναθεωρήσεων στο πλαίσιο και τη δική μας έρευνας και υπάρχει ένας επαρκής έλεγχος και μέτρα παρακολούθησης εντός ε, του WCPFC σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και υποπεριφερειακό επίπεδο ε, περιλαμβάνοντας και το PNA και το εθνικό επίπεδο, το επίπεδο της Παππού Νέα Γουινέας. Υπάρχει η υπηρεσία FFA που έχει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών παρακολούθησης για το WCPFC. Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε το ρόλο των μέτρων διαχείρισης όσον αφορά την τήρηση του Vessel Day Scheme, έτσι όπως έχει καταρτιστεί. Και θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω και έχουν διεξαχθεί κάποιες έρευνες οι οποίες επισημαίνουν το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι διάφορες έρευνες όσον αφορά τη βελτίωση των περαιτέρω μέτρων IUU και επίσης έχει γίνει αναφορά και στις επιπτώσεις ή στην ευθύνη των ε, χωρών ε, σημαίας προέλευση των σκαφών αυτών. Η Παππούα Νέα Γουινέα ε, έχει πολύ αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και παρακολούθηση στην περιοχή αυτή. Και πράγματι είναι από τι καλύτερε στον κόσμο. Το... Όσον αφορά σχέση μεταξύ WCPFC και των υποπεριφερειακών ομάδων, θα πρέπει να πούμε ότι το FFA είναι υπεύθυνο για τις οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των χωρών και δερμέζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των χωρών αυτών για τις διαπραγματεύσεις, το οποίο η Παππού Νέα Γουινέα παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εκπόνηση μέτρων διαχείρισης και διατήρησης. Ε, περιλαμβάνει το Vessel Day Scheme, observer coverage and full catch Τήρηση της κάλυψης κλπ. Και όλα αυτά έχουν ε, αναγνωριστεί ε, μέσω επιστοπίσεων που δείχνουν τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων όσον αφορά την επίτευξη μιας συνένευξης στο επίπεδο της Παππούας Νέας Γουενέας. Τώρα, τα βασικά αποτελέσματα είναι ότι η WCPFC αντιμετωπίζει κάποιες ξεκάθαρες προκλήσεις μεν, αλλά έχουν υπάρξει σημαντικά ωφέλη όσον αφορά την διαχείριση και τα ευεργετικά ωφέλη θα συνεχίσουν. Τα προβλήματα στο επίπεδο αυτό ε, έχουν προκληθεί από μια έλλειψη συμβατότητας όσον αφορά τα μέτρα αυτά, όσον αφορά το πλήρε φάσμα τη αλλίευση. και η Παππούα Νέα Γουινέα συνέβαλε σημαντικά όσον αφορά αυτά τα επίπεδα συμβατότητας, αλλά από την άλλη ε, και από την άλλη έχει καθιερώσει αποτελεσματικά μέτρα ε, και όπως σας είπα το 80% των αλληλευμάτων προέρχονται από αυτή την περιοχή και μέσα αυτών των αποτελεσματικών μέτρων έχουν επηρεάσει σημαντικά την, ε, το επίπεδο, την κατάσταση αφορά της, το επίπεδο λήψη αποφάσεων για μια βιώσιμη αλία στο μέλλον. Έχουμε ακόμη πέντε λεφτά για να δούμε πολύ γρήγορα τις υπόλοιπες διαφάνειες. Όσον αφορά το περιβάλλον, κάποιες ιδέες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μία αρχή διακυβέρνησης και τεχνικά υπεύθυνη και διότι υπάρχουν οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι. Παρ' όλα αυτά, εντοπίσαμε κάποιους κινδύνους εξαιρία της πολιτικοποίησης κάποιων αρχών και δεδομένου ότι το ανώτατο επιτρεπόμενος όγκος αλλιεύματος πολλές ε, φορές, αλλά και τα τελευταία χρόνια, από τότε που εγκρίθηκε το 1980. Τόσο αναφορά το IUU, πρέπει να πω ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δούμε τις αδυναμίες στην χώρα αυτή λαμβάνοντας υπόψη σε ποια περιοχή βρίσκεται, διότι το σύστημα της ε, γενικότερα όσον αφορά την Ελία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Τρεις είναι οι κύριες ιδέες. Πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να δούμε ε, όσον αφορά τη διαχείριση της αλληλεγγύας τις ε, αρνητικές επιπτώσεις. υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την υπεραλίευση, λαμβάνεται τα κατάλληλα μέτρα. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, αηφορία των ε, πόρων των ελιευτικών, πρέπει να πούμε ότι μάλλον είναι θετικά τα πράγματα. Οτιδήποτε προωθεί την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και τους κανόνες ασφαλείας ε, ακολουθείται. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη αξιολόγηση των επιπτώσεων της αλληλευτικής αυτής δραστηριότητα της Παπουαζίας Νέας Γουινέας όσον αφορά την ε, αλληλεία. Υπάρχουν ε, προβλήματα και αδυναμίες όσον αφορά τον ε, έλεγχο και την εποπτεία. Τελικά, ποιο είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις. Η συνθήκες που αφορούν την ε, εργασία και τους μισθούς που καταβάλλονται ευθυγραμμίζονται με τις εθνικούς κανονισμούς που ισχύουν. Ε, δεν είναι πολύ μεγάλη η μισθή. Το κύριο θέμα είναι οι άδειε μητρότητος. Απ' την άλλη, η βιομηχανία του τόνου στη χώρα αυτή θεωρεί ότι δημιουργεί αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις που εξηγούνται εν μέρη εξαιτία των παραδόσεων και την άλλη δεδομένου ότι οι ενεχόμενοι όλοι δεν δίνουν τι απαραίτητε συνθήκες. Πρέπει επίσης να σας πω ότι για λόγους παράδοσης και κουλτούρας ε, οι γεωκτήμονες και αυτοί οι οποίοι κατέχουν τις διάφορες εκτάσεις πρέπει να έχουν κατά κάποιο τρόπο πρώτη μισιακή συμφωνία με αυτούς που εκμεταλλεύονται ε, το προϊόν αυτό και τελικά πρέπει να πω ότι κυρίως στην περιοχή του Μαντάγκ ε, υπάρχουν αιτιάσεις ότι αυτή η βιομηχανία έχει οδηγήσει σε μια έξαρση της πορνείας. Δεν υπάρχουν όμως αρκετά στοιχεία. Ε, η εξέβρεση ε, αλλιευτικών πόρων για, για το συγκεκριμένο ψαριακό δεν έχει οδηγήσει αλλαγές των ε, κοινωνικών επιπτώσεων και μπορεί το θέμα αυτό της προμήθειας ελευτικών πόρων να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι παραμένουν οι βασικοί μισθοί αρκετά χαμηλοί και θα πρέπει Επίσης να ληφθεί υπόψη από την βιομηχανία, η κουλτούρα και η παράδοση η τοπική για να μπορέσει να υποστηριχθεί η, τοπική, η οικονομική ε, ανάπτυξη της περιοχής. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους. Λέει Πρόεδρος, πριν να δώσω, να δώσω το λόγο στον ε, πρόεδρο της ίντα και στους συναδέλφους, θα καλέσω και τον David Μάρτιν, εισηγητή εκ μέρους της ίντα. Αρχίζουμε με τον κύριο Βιτάλ Μορέιρα. Για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είμαι εδώ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Συμμερίζομαι πλήρως την ιδέα ότι όντω θα πρέπει να συνεργαζόμαστε για θέματα κοινά και κοινή ευθύνη, μεταξύ των οποίων αυτό το οποίο συζητείτε σήμερα. Οι περισσότερες συμφωνίες, ε, οι δικέ μας συμπεριλαμβάνουν ε, μία διάσταση ε, όσον αφορά την αλία. Κατά συνέπεια, πρέπει να σας πω ότι και εγώ και η Επιτροπή μου, εάν πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι το θετικό για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συνεργαστεί με σας. Έχουμε εδώ τον συνάδελφο David Martin, ο οποίος ήταν εισηγητής στην Επιτροπή μας για αυτό το φάκελο. Ίσως θέλει και εκείνος να πει κάτι για την Επιτροπή σας για την μελέτη σας. Σας ευχαριστούμε που αναθέσατε αυτή τη μελέτη στους εμπειρογνώμενες. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούμε έτσι να κρίνουμε την κατάσταση και τις εξελίξεις ενδεχομένως σε τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα με τους συναδέλφους την κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της έκθεσης αυτή τους εμπειρογνώμενες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή επέκρινε πολύ η Επιτροπή μας. Η μελέτη που είχε γίνει από την Γενική Διεύθυνση Trade για την ε, παραβίαση των κανόνων ε, ε, που ισχύουν για την, τους κανόνων καταγωγής για την Παπουαζία. Αυτό είπαμε ότι έχει επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή μηχανία. Δεν επιμένω, συγκεκριμένη περίπτωση, διότι τα πάντα μπορούν να έχουν επίπτωση και υπάρχουν άλλες αναπτυξιακές πτυχές οι οποίες δεν είναι σημαίνουσες. Εδώ όμως απεδείχθη ότι μπορούμε να έχουμε επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και πιστεύω ότι αυτό αναλύεται πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι ελέγχθη ότι η μελέτη αυτή είναι περιγραφική, δεν είναι ποσοτική και εδώ σύμφωνα με τα πρότυπα που παρουσιάστηκαν βλέπουμε πώς μπορούν όλα αυτά τα θέματα να έχουν επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κατά συνέπεια επισημένονται πράγματα τα οποία κάποια στιγμή στο παρελθόν είχαμε πει. Δηλαδή ότι δεν έχει γίνει πολύ σωστά αυτή η μελέτη επιπτώσεων από τη Γενική Διεύθυνση Trade. Δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την Γενική Διεύθυνση Trade και υποφελούμε με, από την παρουσία των εμπειρογνώμων και του κυρίου Μορέιρα είναι κάτι το οποίο αναλύεται πολύ ενδιαφέρον στη μελέτη αυτή. Πολλές φορές στο εμπόριο τα θέματα της αλίας και κυρίως αυτά που αφορούν τον τόνο την χάνουν μια πολύ επιφανειακής μετυχείρισης. Η, δεν το λέγω για την ίντα, το λέγω για τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Γενική Διεύθυνση Trade. Και με μεγάλη σαφήνεια αποδεικνύει η μελέτη στην περίπτωση της Παπουαζίας Νέας γυναίκα, ότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό γιατί είναι πολύ μακριά, δεδομένου ότι κοστίζει η ηλεκτροδότηση, διότι δεν υπάρχουν ε, αρκετοί δάτινοι πόροι. Το κόστος λοιπόν παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό. Δεν είναι λοιπόν ανταγωνιστική, παρά μόνον η παποζία Νέα Γινέα, διότι υπάρχει απόκληση από τους ε, κανόνες προέλευσης. Και έτσι βλέπουμε ότι ενώ στο παρελθόν έκανε εξαγωγές προς άλλες χώρες και υπήρους, τώρα έχει μόνο τράτο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Παπουασία Νέα Εάν λοιπόν στο μέλλον το Βιετνάμ, και εκεί νομίζω ότι αρχίζουν διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, η περιοχή του ΑΣΕΑΝ, αν λοιπόν γίνουν τέτοιου είδους, συναυτούν τέτοιου είδους συμφωνίες και έχουμε ανταγωνιστικές χώρες, Εάν ε, τελωνιακοί δεσμοί είναι μηδενικοί ή ε, ισχύουν και εκεί οι αποκλήσεις, τη στιγμή λοιπόν που δεν θα υπάρχει και για εκείνους ε, τελωνιακός δεν θα έχει να κάνει τίποτε στην ε, περίπτωση αυτή με τον τόνο η Παπποζία Νέα Γουινέα δεδομένου ότι οι χώρες αυτές θα μας πλημμυρίσουν με παρέμφερη προϊόντα, με τόνο δηλαδή. Οποιαδήποτε λοιπόν αλλαγή κάνουμε, σίγουρα θα έχει επιπτώσεις, το αναφέρω ως παράδειγμα, για την Παπουαζία Νέα Γουινέα. Αυτοί που ασχολούνται με το εμπόριο, και το λέω πολλές φορές, ότι κάνουμε εμπορικές ε, συμφωνίες ή πράξεις, ελαφρά την καρδία, χωρίς να δούμε τι γίνεται εν βάθη, καταλήγουν σε τέτοιες καταστάσεις. Εδώ εμφανίζεται και ο Ισημερινός εάν αρχίσουν να έχουμε αποκλήσεις των κανόνων προέλευσης και με τον Ισημερινό και εκεί δεν θα έχουμε ανταγωνισμό. Το λέγω αυτό για τα μελλοντικά θέματα τα οποία αφορούν τις διαπραγματεύσεις στην Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα μπορούσαν να υπάρχουν με την σύναψη συμφωνιών με αυτές τις χώρες για την αγορά του τόνου. Τώρα, θα περάσω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μου φαίνεται πιο σημαντικό, πολύ σημαντικό θα έλεγα μάλιστα, και εγώ διαφοροποιούμε από αυτά τα οποία ελέγχθησαν στη μελέτη όσον αφορά τις επιπτώσεις περιβαλλοντικές. Εδώ και κάποιες ώρες παρακολουθώ ε, τις εργασίες αυτής της Επιτροπής Western Pacific. Ξέρουμε περί τίνος ομιλούμε, ξέρουμε ότι όντως πρόκειται για μια ε, επιτροπή για ένα ίδρυμα ατυπική δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό με αποκλειστικές, ε, με ύδατα που βρίσκονται σε αποκλειστικά οικονομικές ζώνες και όχι με ζώνες ανοιχτής θαλάσσης, αφορούνται όντως χώρες οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες αλλά πρόκειται για μια περιφερειακή οργάνωση αλληλεία, η οποία είναι σημαντική. Υπάρχουν θέματα τα οποία εγώ δεν κατανοώ πάρα πολύ καλά για το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μοναδικό μέρο που υπάρχει για τον έλεγχο τη ε, ε, δυναμικότητα ε, τι είναι μείωση τη δυναμικότητα αλλίευση σε ποσοστό 30% πράγμα το οποίο δεν επιτεύχθηκε. Διότι μειώθηκε και ο λευτικός στόλος, τις προβλέψεις που κάνετε εσείς για ε, τα αλλιεύματα στην Γοηναία Νέα Παπαζία από 90.000 τόνους περάτε σε 200.000 τόνους, πράγμα που είναι σημαντικό αύξηση των ε, αλλιευμάτων. Και εδώ μιλάμε για μείωση τη δυναμικότητας παρά για αύξηση. Άρα, ό,τι και να λέγεται, πέρσι είχαμε αύξηση 18% για τα Vessel Day Scheme στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Δεν υπάρχει έλεγχος του Vessel Day Scheme ή ελάχιστος έλεγχος, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και ούτε καν εφαρμόζεται αυτό στα ανοιχτά ύδατα, στην ανοιχτή θάλασσα που είναι εντός αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτό το Vessel Day Scheme. Κάθε χρόνο ε, ορίζεται ένας νέος αριθμός, ανώτερος αριθμός ημερών που επιτρέπεται η αλία, γιατί κάθε χρόνο ξεπερνιέται αυτό που έχει οριστεί, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος. Άρα δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό. Όσον αφορά τις ε, ζώνες ανοιχτών, ανοιχτής θάλασσας εξαιρούνται από οποιαδήποτε κανονισμό και αυτό είναι ενάντιο πως αυτό το οποίο γίνεται ε, για την αλία του τόνου παντού εντός των αλιευτικών αποκλειστικών ζωνών. Άρα κυρίαρχο κράτο, η Παπόζια Νέα κάνει ό,τι θέλει ακόμη και σε διεθνή ύδατα. Και δεν σέβεται τίποτα αν τη συμφέρει. Και βεβαίω δεν θα μιλήσω καθόλου και για τα τσάρτερ, για τα αναβλωμένα σκάφη τα οποία έχει. Έχει 40 αναβλωμένα σκάφη και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στη Western. Δηλαδή, η ναύλωση πέρσι έγινε με μεγάλη ε, είπαμε για την περσινές ναυλώσεις, ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν ώρες-ώρες τα φορτώματα αυτά. Εσείς είπατε ότι περνούν από τη μεταπητική βιομηχανία. Όντως υπάρχει μία, ε, ένα υπουργείο που συνεχίζει να ασχολείται με αυτά τα θέματα, αλλά δεν ταξιδεύουν τη μεταποιητικη υπάλληλοι και τυχαία εκεί που είναι το υπουργείο βρίσκονται και όλοι οι υπάλληλοι, δεν μετακινούνται, στέλνουν κάποιες εκθέσεις αλλά κανένα δεν πάει επί τόπου να εξακριβώσει περί τίνο πρόκειται και να κάνει διαπιστώσει. Εκπλήσαμε λοιπόν που και εσείς, ε, όπως λέτε, υπάρχει παράνομη ε, αλία. Το θέμα αυτό είναι, όπω ξέρετε, δύσκολο αμφιλεγόμενο και δύσκολα μπορούμε να βρούμε λύση. Κατά συνέπεια συνεχίζω να λέω ότι τα μέτρα για το περιβάλλον και οι επιπτώσεις που όλα αυτά μπορούν να έχουν στο μέλλον αυτή τη στιγμή είναι Κάτι που μου προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά. Και εσείς συνάγετε το συμπέρασμα ότι η Κίνα, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ και οι χώρες που αναπτύσσουν παρεμφέρει βιομηχανία, γιατί πηγαίνουν εκεί. Για την πρώτη ύλη. Εσείς οι ίδιοι το λέτε, ότι το κόστος παραγωγής είναι, ε, διαμορφώνεται με 61% κόστος της πρώτης ύλης και τα υπόλοιπα είναι άλλα κόστη. Οπωσδήποτε είστε σε μια περιοχή που είναι από τις πιο πλούσιες σε τόνο, αλλά ε, η, ανηφορία, αηφορία τι κάνει, τη λαμβάνετε υπόψη. Επίσης, νομίζω ότι... Αυτά ήταν τα κυρία σημεία που ήθελα να θίξω. Δεν έχω να πω ότι περισσότερο. Τέλος πάντων, το άπα όλα, τα άπα όλα και μακριγώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Φράγκο, κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτή την επιτροπή. Θα είμαι σύντομο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω του συντάκτε τη μελέτη. Είναι πάντα καλό να έχουμε κάποιο έγγραφο βασιστό που μπορούμε να συζητήσουμε. Όπω γνωρίζετε, όταν αυτή η συμφωνία Σύμπραξη ε, ε, παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο. Εγώ είπα να την υποστηρίξουν για αναπτυξιακού λόγου και πιστεύω ότι η μελέτη έχει ενισχύσει τι ε, απόψει μου ότι πρόκειται για μια καλή αναπτυξιακή ευκαιρία για την Παππού Ανέγουινέα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε με τι χώρα έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε μια χώρα που είναι πολύ μακριά από τις κύριες αγορές, ακόμη και από την Αυστραλία. Είναι πολύ δύσκολο για αυτήν να, να παράγει τα μηχανικά προϊόντα. Βασίζεται στην Αλία ω ένα από τα κυριότερα προϊόντα της έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας, ε, ιδίως ε, μεταξύ των γυναικών και έχει υποφέρει τελευταία από πολιτική αστάθεια. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας ε, είναι καλή είδηση και από ό,τι ακούμε από τους συντάκτες της μελέτης κάποιες ελπίδες ευδόθηκαν. Όπω φαίνεται, υπάρχουν αυξημένε επενδύσει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης. και αυτό εκπλήρει έναν από του ανεπτυξιακού μα στόχου να προσθέτουν αξία στα προϊόντα του και η, η Παπώνια Γουινέα κονσερβοποιεί τόνο εντό του εδάφου τη και αυτό δημιουργεί νέες πηγές οδήματος μέσω της ε, προμήθειας ε, προϊόντων αλληλευτικών σε άλλες χώρες το οποίο επηρεάζει πολύ θετικά τη χώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι στο σύνολό του αυτέ οι ειδήσει που μαθαίνουμε ότι η οικονομία τη Παπασδανή Γουινέα βελτιώνεται είναι πολύ καλή. Και φυσικά εκφράζονται κάποιε ανησυχίε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Αυτό που θα ήθελα να πω. Ε, επειδή υπήρξε αύξηση των εκφορτώσεων ψαριών στην Παπαναγουενέα, αυτό δεν σημαίνει καθαρή αύξηση στα μεταποίηση ψαριών. Ορισμένα ψάρια απλά ήρθαν από άλλες... Α, δεν σημαίνει αύξηση των ελευμένων ψαριών. Ε, κάποια ψάρια προήλθαν από άλλες πηγές. Ε, συνεπώς ε, διαφέρει η ποσότητα αλλιευμένων ψαριών και η ποσότητα εκφορτωμένων ψαριών. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση όσον αφορά το περιβάλλον και το πιο σημαντικό που είπατε και συμφωνώ απόλυτα με αυτό είναι ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα με τις άλλες εμπορικές συμφωνίες ώστε να μην ε, δημιουργήσουμε κάποιο προτιμησιακό καθεστώς για την Παπονέου. Είναι, τις έχουμε δώσει ένα μικρό πλεονέκτημα, αλλά δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε από την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ τα ωφέλη που έχουν ήδη. Ε, ε, θα πρέπει να προσέξουμε όμω με την ΠΕΠΑ ώστε να μην βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Θα πρέπει να προσέχουμε πολύ όσον αφορά το προτιμησιακό καθεστώ. Το ίδιο είχε γίνει και με τη Συμφωνία Λευκή Σύμπραξη στην Καραϊβική. Είχαμε δώσει πολύ καλό προτιμησιακό καθεστώ για τι μπανάνε και μετά όταν ε, κάναμε εμπορικέ διαπραγματεύσει με την Κεντρική Αμερική. Ε, υπήρχε κάποιο θέμα με την Καραϊβική. Δεν θέλουμε λοιπόν να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος και στην Αλία. Αλλά σήμερα έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία ε, λειτουργεί και θα πρέπει να συνεχίσουμε φροντίζοντας να προστατεύονται και τα υπόλοιπα ζητήματα, το περιβαλλοντικό ζήτημα σε αυτό το μέρος του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάρτιν. Ναι, υπήρχε πράγματι αυτή η απογοήτευση για τους Ευρωπαίους παραγωγούς όσον αφορά την μπανάνα, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς από τα Κανάρια. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους ε, συντάκτες της έκθεσης. Ναι, Ωραία. Ένα από τα θέματα τα οποία θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπε η κυρία Φράγκα είναι η ευξενόμενη ζήτηση από τις βιομηχανίες του Παππούα Νέα Γουινέα. Υπάρχει μια ποικιλία όσον αφορά τα λεύματα. Οι, αυτοί που κάνουν κονσέρβες παίρνουν μια, ένα πολύ μικρό μερίδιο από τα λεύματα. Και ε, δεν σημαίνει ότι συνεπάγεται ακριβώς μια αύξηση των ε, αλευμάτων ε, που εφόσον διατηρείται το Vessel Day Scheme. Απλώς υπάρχει μια καλύτερη οικονομική αξιοποίηση όσον αφορά αυτά τα λεύματα στην Παπουασία Νέα Γουινέα. Και εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Φράγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά την ε, μείωση της συνεισιμότητας των αλευμάτων κατά 30%. Αυτό αφορά κυρίως για τον, ε, τον μεγαλόφθαλμο τόνο και τον ε, κυτρινοπτερίγιο, κυτρινο, κυτρινόπτερο συγγνώμη, τόνο. Αλλά η πλειονότητα των αλευμάτων είναι παλαμίδες και αυτοί δεν αξιοποιούνται Τώρα, το θέμα, το θέμα των υδάτων αυτών του αρχιπελάγους είναι ένα θέμα, ιδιαίτερα σε αφορά την Παπουασία Νέα Γουινέα. Εδώ είναι περίπου το 15% των αλευμάτων προέρχεται από την Παπασία Νέα Γουινέα και πράγματι υπάρχει μια ανησυχία εδώ, αλλά ο αντίκτυπος είναι σχετικά περιορισμένος όσον αφορά το σύνολο των ελευμάτων από τα ύδατα της Παπουασίας Νέας Γουινέας. Επίσης υπάρχουν κάποια θέματα όσον αφορά τις ημέρες αλίευσης και την υπεραλίευση. Ε, πράγματι έχει διαπιστωθεί μια αύξηση στα αλιεύματα και θα ήθελα να αναφερθώ στις έρευνες που αναφέρουν κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα νέο ή τριών ετών ε, και έχουν, το οποίο έχει, έχει δεχθεί κάποιες αλλοιώσεις και θα υπάρξουν περιττέρω αλλοιώσεις. Υπάρχουν κάποια σχετικά σχόλια. Τώρα, η αξιολόγηση που έχει γίνει από τις εκθέσεις είναι όσον αφορά την αλληλευτική ικανότητα είναι ότι οι αρχές της Παπουασίας ε, Νέας Γουινέας είναι σε θέση να διαχειριστούν το θέμα αυτό. Στην έρευνα ε, διατυπώθηκε μία επιφύλαξη όσον αφορά τη διαχειρισιμότητα ε, και σε σχέση με μία περιβαλλοντική πτυχή που αφορά τη μόλυνση από τις βιομηχανίες. Και υπό την έννοια αυτή, ε, όλα τα, τα όλες οι βιομηχανίες είχαν καλά συστήματα καθαρισμού αλλά ίσως η διενεργούμενη έλεγχη δεν ήταν τόσο συχνή όσο θα θέλαμε. Εν γέννη όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση των αποβλήτων της ε, βιομηχανίας ήταν αρκετά αρκεί στην Παπουασία Νέα Γουινέα ε, όσον αφορά κυρίως τα, την παραγωγή φιλέτων. Στα 60% έχουμε ε, παρόλο το 60% ε, έχουμε 40% το οποίο θα πρέπει κάπως ε, να επεξεργαστεί ως απόβλητο. Ε, είναι, μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόλογο προϊόν το οποίο να εξαχθεί, το οποίο να είναι κατάλληλο προς βρώση. Τώρα, όσον αφορά την βιωσιμότητα, παρόλο που έχει γίνει αναφορά στην αλήψη της παλαμίδας, η οποία δεν έχει γίνει αντικείμενο επαρκούς εκμετάλλευσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια ε, συστήματα, κάποιες προβλέψεις συστήματα μακροπρόθεσμης ε, διαχείρισης σε σχέση με τα μέτρα διατήρησης τα οποία έχουν ένα αρκετά καινοτόμο χαρακτήρα κυρίως για την περιοχή αυτή αλλά και σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο. Ωραία λοιπόν, αν δεν υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση, η κυρία Φράγα. Πριν να ξεχάσω θα πω το εξής. Προσπαθώντας να καταπολεμήσουμε την παράμονη αλληλεία υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το Port State Measure και το Catch Documentation Scheme. Το λέει η ΦΑΟ. Το πρώτο, το Catch Documentation Scheme, δεν ανταποκρίνεται, αν θέλετε, με τους κανόνες, τους κοινοτικούς, όσον αφορά την παράνομη αλληλεία. Τώρα, για το δεύτερο θέμα που ανέφερα. Τα δύο χρόνια που είμαι εγώ παρατηρητήρια στη Western, ζητώ να τεθεί επιτέδιον αυτός του Port State Measures και καμία από αυτές τις χώρες, και άλλες, και άλλες, όπως η Ιαπωνία που δεν θέλει να εφαρμόσει, καμία χώρα δεν θέλει να τα βάλει κάτω για να ελέγξει τα πράγματα. Άρα, επιτρέψτε μου να πω ότι η παράνομη αλληλεία είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και ένα από τα στοιχεία που υπάρχουν στο άρθρο 6 του πρωτοκόλου 2 της συμφωνίας λέγει ότι η συνεργασία πρέπει να υπάρχει μεταξύ της χώρας αυτής και των υπολείπων για θέματα παρανομίας. Και ε, δεν έχει γίνει τίποτα. Και εδώ θέλω να αναγνωριστεί το εξή. Η υποποζία Νέα Γουινέα, γιατί ε, θέλω να είμαι αντικειμενική, κάνει προσπάθειε να βελτιωθεί χάρη στι προσπάθειε που καταβάλει και η Αυστραλία και για πολιτικού λόγου. Πολύ καλό μου φαίνεται αυτό. Και νομίζω ότι όλοι οι ανεπτυγμένες χώρες εμείς έχουμε καθήκον να βοηθήσουμε τους άλλους να απτυχθούν. Χάρη λοιπόν στις επικρίσεις που κάνουμε και εκείνοι προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση. Σωστό, σωστό μου φαίνεται αυτό, ο σωστός δρόμος. Αλλά μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να γίνουν και να ξέρω ότι αυτά τα θέματα της παράμεσα αλληλείας είναι θεμελιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Εάν όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εισηγητές της μελέτης αυτής και όλους εσάς. Όπως είπα και στην αρχή, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο Μορέιρα και τον κύριο Μάρτιν που είναι παρόντες. Είναι η πρώτη φορά που είσαστε εδώ, σας καλέσαμε, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι τελευταία. Έξι υπακούεται, λέει ο κύριος Μορέιρα. Πού τώρα εδώ. Ε... Continuamos con Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 16. Τροποποίηση του κανονισμού 812 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεπίπτοντα αλλιεύματα και το ειδών κατά την και για την τροποποίηση του κανονισμού 88 κάθετος 98. Σήμερα η Επιτροπή θα μας παρουσιάσει την πρότασή της και από μεριά μα εισηγητή είναι ο κύριο Ρωμέβα. Η Κομισιόν λοιπόν έχει το λόγο για να μα παρουσιάσει την πρότασή τη. Nombre de la Comisión, señor Rian. Κύριος εκ μέρους της Κομισιόν. Όχι, κάποιος άλλος. Όποιος θέλει. Ναι, αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο αργά. Ωραία και πάλι. Αυτή η πρόταση αφορά τον, ε, μια ρύθμιση όσον αφορά το, ε, σε ευθυγράμμιση της, με το πνεύμα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σχετίζεται με τα όσα συζήτησαμε σήμερα το πρωί για την, τον κανονισμό για τα χέλια και αναφέρεται στις αρμοδιότητες που δίδονται στην Επιτροπή όσον αφορά τις ε, κατουσιοδότηση και τις εκτελεστικές ε, πράξεις και προτείνουμε η Συμφωνία να μπορεί να υιοθετήσει ε, πράξη πράξης όσον αφορά την τροποποίηση ορισμένων τμήματων του κανονισμού που αφορά, αφορούν τους όρους χρήσεως ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών όπως ε, ορίζονται στο παράτημα όταν υπάρχει αυτή η ανάγκη ούτως ώστε να υπάρξει τεχνική πρόοδος. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα δίδονται στην Επιτροπή ούτως ώστε να ε, καταπιέζονται οι αιτήσεις εκθέσει σύμφωνα με το άρθρο 8. Ο κανονισμός δεν αφορά με πιο εκτεταμένη αναθεώρηση του κανονισμού. Θα το κάνω πολύ απλά σε σχέση με το τι προγραμματίζει η Επιτροπή για την αναθεώρηση. Ήμουν εδώ, έλαβα υπόψη μου τα σχόλια, ωστόσο θα προτιμούσα να δω το ίδιο το κείμενο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, τα οποία θα ήθελα να ελέγξω και θα το κάνω το ταχύτερο δυνατό. Και καταλαβαίνω ότι αυτή η διαδικασία είναι αυτή η οποία έχει καθιερωθεί ούτω ή άλλω. Δεν βλέπω να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σχέση με αυτή την έκθεση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υπάρχει μια γραμμοδότηση κατά μια γνώμη κατά πόσο αυτό είναι παρκές ή όχι. Συγγνώμη, υπάρχει καμία άλλη παρέμβαση, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Εάν όχι, θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα πάμε προς τα πίσω, θα πάμε στο σημείο υπαριθμών 6 δηλαδή σύναψη του πρωτοκόλου αλευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου σχετικά με τον καθορισμό των αλευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή μεταξύ των δύο πλευρών. Η συγκέντρια είναι η κυρία Πατράο Νέβες. Το Κοινοβούλιο αναμένει μια αναθεώρηση εκ μέρους του Συμβουλίου θα συνεχίσουμε λοιπόν τις εργασίες μας για να δούμε κατά πόσο θα οριστεί κάποια ημερομηνία. Και αυτός ο οποίος μπορεί βεβαίως να περιγράψει καλύτερα την κατάσταση είναι η ίδια η συγκήτρια, η κυρία Πατράου, η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Προεδρία και τον συνάδελφο που επέτρεψα να αλλάξει η παρουσίαση της έκθεσης αυτής, δεδομένου ότι δεν μπορούσα να ήμουν χθε παρούσα. Πιστεύω ότι αξίζει αρχίζοντας να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλιεύει από το 1980 στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου. Έχει υπογράψει διάφορες ε, αλληλευτικές συμφωνίες και ήταν στη διαδικασία υπογραφής ενός καινούργιου όταν πέρσι στις 12 Απριλίου έλαβε χώρα ένα πραξικόπημα εκεί. Κατά συνέπεια, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, η μη δημοκρατική κυβέρνηση που επεκράτησε οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην διακοπή των αλληλευτικών δραστηριοτήτων και την απόσυρση του αλληλευτικού μας τόλου από τα ύδατα εκεί. Στη μεταξύ διάστημα η διαδικασία είχε προχωρήσει αρκετά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε εκ μέρους της Κομισιό, η Κομισιό ενέκρινε το πρωτόκολλο στις 5 Ιουνίου 2012 και νομίζω ότι μπορεί να μας παρουσιάσει τις γενικές γραμμές του πρωτοκόλλου αυτού πριν να περάσουμε σε άλλου είδους παρατηρήσεις. Τώρα, όσον αφορά το πρωτόκολλο αυτό, ειδικά που όπως σας είπα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι προβλέπεται μία ετήσια χρηματική ε, καταβολή στη Γουινέα Μπισάου της ε, τάξης του 22,5% με μείωση των διανατοτήτων αλίας. Αυτή η μείωση δεν σημαίνει οπωσδήποτε η απαραίτητος μείωση και των αλλιευμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι αυξήθηκε το ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλουν οι πλειοκτήτες για την αλληλεύση και υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την αλληλεία Εκεί και αύξηση του κόστους που καταβάλουν για να έχουν δικαίωμα αλληλεία οι Σύμφωνα με τι διάφορες πληροφορίε που είχαμε επίσης εκ μέρους της Επιτροπής, έχουμε να κάνουμε με μία χώρα στην οποία οι ελευτικές συμφωνίες με την Αυρεπική Ένωση και είναι αυτή μια τρίτη χώρα όπως ξέρουμε, συνήθως την χάνουν εποπτείας εύκολα. Είναι εύκολο να γίνει λοιπόν αυτός ο έλεγχος εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η παρούσα κατάσταση, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επειδή δεν μπορούν να λιεύσουν τα δικά μας σκάφη, είναι κάτι το οποίο είναι λυπηρό. Αλλά αυτό εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη χώρα αυτή. Τώρα, όσον αφορά το πρωτόκολλο το εν λόγω, διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση ότι στο πρωτόκολλο αυτό υπήρχε ε, αύξηση των δεσμεύσεων για η φόρο αλία. Είδαμε ότι δεν πρόκειται απλώς για απλή μεταφορά χρημάτων για την Γουινέα Μπισάου, αλλά όντως αναπτύσσεται με τη χώρα αυτή μια πραγματική συμφωνία αλλιευτικής σύμπραξης και υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα και συγκεκριμένα στοιχεία που μας οδηγούσαν στο να πούμε ότι αναπτύσσεται ο τομέας αυτό σε θέματα ελέγχου, σε θέματα ανάπτυξης και βοηθειών και επίσης ε, προβλέπεται σύμφωνα με τη συμφωνία ναυτολόγηση τοπικού εργατικού δυναμικού, πράγμα που είναι σημαντικό για την τοπική οικονομία, βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και της κατάρτισης των ε, εργαζομένων εκεί, πράγμα το οποίο έχει ε, μεγάλες και θετικές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό. Όπως ξέρετε η Γουινέα, η Γουινέα Μπισάου είναι από τις πιο φτωχές χώρες και γενικότερα η κατάσταση ήταν πολύ ικανοποιητική, η έλεγχη ε, και η εποπτεία γίνονταν σωστά, υπήρχε παρουσία παρατηρητών επί των αλλιευτικών σκαφών, υπήρχε σύστημα παρακολούθησης δορυφορική, σύστημα ηλεκτρονικής αναφοράς και Όλα αυτά για να μπορέσουν να μην υπάρχουν υποψίες ότι γίνεται η παράνομη και μη ελεγχόμενη αλία. Επίσης, ε, ε, συστάθηκε κοινή επιστημονική επιτροπή που είναι υπεύθυνο για την συλλογή δεδομένων, για τις ετήσιες αξιολογήσεις, για ε, μέτρα ε, που αφορούν τους, την πρώτη ύλη, τους πόρους, διορθωτικές διαδικασίες και μέτρα, ώστε να υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Πρέπει λοιπόν να πω ότι γενικά το πρωτόκολλο αυτό μου φαίνεται ότι ειλικρινά είναι ικανοποιητικό και κάποια μέτρα ακόμη ξεπερνούν το σύνηθες πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται άλλου είδους πρωτόκολλα που έχουμε αναλύσει εδώ με άλλες χώρες. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να τύχουν βελτίωσης, αλλά γενικά Όντως πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα πρωτόκολλο το οποίο είναι σχετικά θετικό. Αρκετά θετικό μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά το κόπημα έχουμε μία παράνομη κυβέρνηση που ηγείται της Γουινέας Μπισάου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στις 2 Ιουνίου, όταν για πρώτη φορά έκανα εδώ την παρουσίαση ή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το πρωτόκολλο αυτό με την Γουινέα Μπισάου, ερώτησα τους συναδέλφους το εξής. Μη πρέπει εμείς ε, στην, να προχωρήσουμε εδώ με την εργασία που κάνουμε στην ε, Επιτροπή Ελίας. Χωρίς να ασχοληθούμε ε, Λαμβάνοντα υπόψη ότι όντω πρέπει να αποκατασταθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες, να ακολουθήσουμε εμεί την τεχνική μα διαδικασία, διότι εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν αξίζει να προχωρήσουμε. Το συζητήσαμε αυτό πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και εγώ ήθελα να ξέρω αν μπορούμε να συνεχίσω, εγώ αν πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά μου ή όχι για αυτό το θέμα αυτό με την επιφύλαξη ότι δεν θα συγκεκριμενοποιήσουμε τίποτε εάν δεν επανέλθει δημοκρατική και συνταγματική τάξη στη Γουινέα Μπισάου. Και όλοι οι συνάδελφοι είπαν ναι, να προχωρήσουμε μέχρι εκεί που είναι δυνατόν στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής μας. Αυτά έγιναν στις 12 Ιουλίου. Αφού επιστρέψαμε τις καλοκαιρινές διακοπές, στις 4 Σεπτεμβρίου Ζήτησα συνάντηση με τον κύριο Μανουέλ Μπέρτ, ε, υπεύθυνο τμήματάρχη της Επιτροπής και με την κυρία Ιζαμπέλ Βιαλό, υπεύθυνη της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ, για, ΜΑΡΕ για το φάκελο αυτό, για να κάνουμε αξιολόγηση της κατάστασης. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στην Επιτροπή Ελίας θεωρήσαμε ότι άξιζε τον κόπο να προχωρήσουμε στα πλαίσια των δυνατήτων και συγχρόνως Πρέπει να πω ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η ίδια με αυτή την οποία είχαμε υιοθετήσει εμείς τον Ιούλιο. Έτσι λοιπόν εγώ προχώρησα βεβαίως με την έκθεσή μου και είχε προβλεφθεί η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών στις 13 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό παρουσίασα εγώ την έκθεσή μου στις 10... Με συγχωρείτε, παρουσίαση της έκθεσης είχε 13 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ίδια ημερομηνία λοιπόν μου είπε η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ ότι δεν μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και ζητήθηκε παράταση για να γνωμοδοτήσει για αυτό το σχέδιο σύστασης. Εμένα με εξέπλησε αυτό, διότι εμείς δεν είχαμε αλλάξει τίποτε. Ε, υποθέτω ότι η Επιτροπή Ντέβερ θεώρησε ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτε, διότι εμείς δεν αλλάξαμε καθόλου τα χρονοδιαγράμματα. Αλλά επειδή δεν υπήρχε πίεση εκ μέρους μας, πίστευα ότι θα μπορούσαμε εύκολα να καταλήξουμε με την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ σε συμφωνία και να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται ώστε να μπορέσει όντως να γδομοδοτήσει. Εμάς δεν μας πίεζει το χρόνος επειδή έτσι έχουν τα πράγματα και αυτό συμφωνήσαμε. Η ΔΕΒΕ θα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή στις 6 Δεκεμβρίου Αυτό συμφωνήσαμε. Για να έχει χρόνο η Ντέβε να κάνει τη δουλειά της. Στο στις 25 Σεπτεμβρίου πήρα κάποιες πληροφορίες ότι όσον αφορά τη διαδικασία είναι απαραίτητο το Συμβούλιο να αποστείλει επίσημο Έτοιμα προσφυγής, ώστε να περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όντως εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις διαδικασίες. Ε, προχώρησα σιγά σιγά, έλεγα πάντα στους ε, διάφορους ενεχόμενους τι κάνω, τα είπα όλα αυτά τα οποία είπα τον Ιούλιο στην Επιτροπή μας και στις αρχές Σεπτεμβρίου τα ξαναείπα και τώρα ενημερώθηκα από τη Γραμματεία μετά από την παρουσίαση της έκθεσης στις 25 Σεπτεμβρίου ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω διότι πρέπει να περιπαίνουμε το θέμα αυτό της ΕΖΗΝ να το παρουσιάσει το Συμβούλιο για να περάσουμε στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Εφόσον λοιπόν έχουν έτσι τα πράγματα και εφόσον αυτό μου είπαν ή οι δήμονες ότι μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο σύστασης μετά από την 6η ε, ε, Δεκεμβρίου. Και αυτό το επίσημο αίτημα του Συμβουλίου έχει σχέση με τη δημοκρατική αποκατάσταση του πολιτεύματος στην Γουινέα Μπουισά. Τι να πω. Εκφράζω τη λύπη μου. Διότι όσοι είχαν αυτή την πληροφορία δεν με ενημέρωσαν έγκαιρα. Διότι εγώ παρουσία στην εκθεσή μου, στην προθεσμία που είχα μπροστά μου και αφού περάσαμε από αυτές τις ε, διαφορετικές ε, στάδια διαδικασίας. Σήμερα ακούσαμε να λέει η Επιτροπή ότι όντως άξιζε τον κόπο να προχωρήσουμε, όσο πιο μακριά δηλαδή, όσο πιο πολύ να προχωρήσουμε, διότι όταν αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Γουινέα Μπισάου, δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και εμεί, βεβαίως ποτέ δεν είχαμε τέτοιου είδου πρόθεση. Δεν είχαμε πρόθεση να κάνουμε το αντίθετο. Ε, λοιπόν, είναι έτοιμη η έκθεση. Εγώ περιμένω η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ να γνωμοδοτήσει και όπως εξήγησε, δεν θα κάνουμε τίποτε εάν δεν αποκατασταθεί η δημοκρατία στη Γουινέα Μπισάου. Όπως πολλοί γνωρίζουν, η Πορτογαλία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί το θέμα αυτό, δεδομένου ότι η Γουινέα Μπισάου έχει με μας προνομιακές σχέσεις, δεδομένου ότι ήταν μια πρώην πορτογαλική απικία, καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Μπορώ Επίσης, να πω σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την όλη διαδικασία ότι περίπου πριν από 10 μέρες ο πρώην πρόεδρος της Γουινέα ε, Μπισάου συνάντησε τον νυν πρόεδρο, τον πραξικοβηματία δηλαδή, συναντήθηκαν στον Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ για να δουν πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουν στις ε, πολιτικές ε, σχέσεις ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη. Και πιστεύω ότι είναι ε, παράξενο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εκτός της χώρας να συναντώνται και να μιλάνε μεταξύ τους ένας ε, πρώην πρόεδρος και αυτός ο οποίος πραξικοπηματίας του έχει φάει τη θέση. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά ίσως υπάρχει μια κάποια βούληση να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη Γουενέα. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας έκθεση, δεν μπορώ να πω να προσθέσω τίποτα άλλο και δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Señora ναι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πράγματι, πρόκειται για ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει ανασταλεί μετά από το πραξικόπημα το πρωτόκολλο αυτό είχε γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση με τις νόμιμες αρχές πριν από το πραξικόπημα στη Γουινέα Μπισάου. Το πραξικόπημα έγινε τον Απρίλιο. Το Συμβούλιο έλαβε κάποιες άλλες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την παρήτητα της κατάστασης για τα άτομα εκείνα τα οποία απείλησαν τη σταθερότητα και την ειρήνευση στην περιοχή αυτή και αποφάσισε την αναστολή της αναπτυξιακής βοήθειας προς τη Γουινέα Μπουισάου και βεβαίως ε, έδωσε προτεραιότητα στην ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης η Επιτροπή απίφθινε μία σύσταση ε, να Λέγοντα ότι αν δεν αποκατασταθούν ε, οι συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο στην ε, Γουινέα Μπισάου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φράγα έχει το λόγο. Εγώ επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, αλλά ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι κρίμα από την λευτική άποψη, από την πολιτική άποψη. Εγώ βεβαίως θα μιλήσω από την άποψη της ε, αλίας. Από, τα, από τρεις ε, συμφωνίες αλληλευτικής ε, σύμπραξης που είναι το Μαρόκο, η Γουινέα Μπισάο και η Μαυριτανία. Στην Μαυριτανία έπαυσε για τα προβλήματα που είχαν και, και κανείς δεν λέει πλέον στα τα αυτά. Ε, στο Μαρόκο ακούσατε σήμερα ότι επίσης έχει ανασταλεί η συμφωνία ε, και το θέμα όσον αφορά τη Γουινέα Μπισάου, για, άλλα λόγα, ε, για άλλους λόγους επίσης υπάρχει αναστολή. Μιλούμε για έναν στόλο ο οποίος δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα στην περιοχή, γιατί πρόκειται, για ειδικέ συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης. Και βεβαίως αφορά θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, θα ήθελα να πω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία στην Επιτροπή, αλλά όχι στην Ολομέλεια. Μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή ε, σε σχέση με την... όπως έγινε με τη Χιλή όπου έγινε και τον, το, την αλία του Ξηφία εκεί και έγινε η σχετική ψηφοφορία. Μπορούμε να, ε, μπορεί να διεξαχθεί λοιπόν η ψηφοφορία και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεγάλο βαθμό αναμένοντας να εξομαλυνθεί η πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή ούτε ώστε να μπορέσουμε ένα, ο στόλος μας να έχει κάποια πρόσβαση σε αυτά τα ελευτικά ύδατα, γιατί πραγματικά όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο κόστος και οικονομικές επιπτώσεις. Και στο τέλος της περίοδου προγραμματισμού ε, δεν θα υπάρχουν καθόλου χρήματα. Και όλα αυτά έχουν δραματικές υποπτώσεις για το τομέα. Γιατί ο ίδιος ο τομέας βεβαίως δεν είναι υπεύθυνος στις πολιτικές εξελίξεις, αλλά υποφέρει από τις επιπτώσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε κάπως ευέλικτοι αναμένοντας να εξομεληθεί και να υπάρξει δημοκρατική μετάβαση στη χώρα. Εξ ονόματος της συναδέλφου Σαββέλα Λοβίν ε, μιλώ, που είναι σκιώδη. Σήμερα όμως δεν μπορούσε να είναι εδώ, γι' αυτό Μιλάω εγώ εκ μέρους της. Διαβάζοντας την πρόταση έκθεσης και βλέποντας πώς έχει η κατάσταση αυτή και ακούγοντας την εισηγητρία, έχω μεγάλες αμφιβολίες. Δηλαδή, παρακολουθούμε τι, συμβαίνει από πολιτικής πρόταση, αλλά προς τα πού θα τραβήξουν οι εξελίξεις δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν μάλλον υπέρ του να ακολουθήσουμε τη γραμμή του Συμβουλίου, να σταματήσουμε τη διαδικασία διότι φοβούμε ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εδώ, ό,τι ψηφί, ό,τι συζητήσουμε δεν θα έχει καμία χρησιμότητα τη στιγμή που θα ψηφίσουμε ή θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν πιο λογικό να περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΖΗΝ του Συμβουλίου για να ξέρουμε βασικά ε, βάσει ποιων στοιχείων μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αβεβαιότητες όσον αφορά την κατάσταση και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα δεν χρειάζεται να αναλώσουμε τους πόρους μας εδώ και να δουλέψουμε για ένα θέμα που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Η δική μας η ομάδα λοιπόν είναι αντίθετη πριν να γίνει οτιδήποτε που θα μας οδηγήσει στο να έχουμε περισσότερη ε, γνώση του τι ακριβώς σημαίνει. Κύριε Στόρμπεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αν υπάρχει μία χώρα που χρειάζεται δημοκρατική ανάπτυξη, αυτή είναι σίγουρα η Γουινέα Μπισάου. Εάν δούμε την ιστορία της των τελευταίων 50 ετών, η ιστορία της είναι πραγματικά θλιβερή με πραξικοπήματα και φόνους και σφαγές ε, μετά από το φόνο του Καμπράλ και η ιστορία της γενικά δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν θετικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Όταν διαβάζει κανείς τις ειδήσει αυτή τη στιγμή, και στην τοποθεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ Νέα Μπισάου χαρακτηρίζεται ως κέντρο λαθρεμπορίας ναρκωτικών, για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και τα πράγματα επιδεινώνονται μετά από το πραξικόπημα. Δεν είναι απλά ένα πρόβλημα δημοκρατίας, υπάρχει ένα πιο βαθύ πρόβλημα για το πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Υπό αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνω τις απόψεις, την άποψη που προωθείται εδώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε το ταχύτερο δυνατόν. Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθούμε τώρα. Σίγουρα να κινηθούμε τώρα. Πρέπει σίγουρα να αναβάλουμε οποιαδήποτε δράση για αυτό το ζήτημα μέχρι να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Θέλει να πει κάτι η Κομισιόν από αυτού του θέματος. Γεια σας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Εμμανουέλ Μπέρκ που δεν μπόρεσε να παραστεί απόψε. Η Κομισιόν θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Πατρονέβες για την προπασκευαστική της δουλειά σε αυτό το φάκελο. και όλα αυτά παρά την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα. Καθώς η κυρία Μπατρονέου εξήγησε ιστορικά, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία μας με την Κινέα ήταν μια χαρά. Αυτό επέτρεψε ε, μια ομαλή διαπραγμάτευση στα τέλη του 2011 αρχές του 2012 που κατέληξε στη μονογραφή του νέου πρωτοκόλλου το Φεβρουάριο του 2012 υπό ικανοποιητικές συνθήκες. Δυστυχώς ε, στη συνέχεια τον Απρίλιο έλαβε χώρα το πραξικόπημα το οποίο ξανέθεσε τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Από τον Απρίλιο λοιπόν ε, συστήσαμε στο στόλο να εγκαταλείψει τα ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακόψει οποιαδήποτε σχέση με τη Γουινέα Μπισάου. Έτσι λοιπόν το προηγούμενο πρωτόκολλο έληξε στι 15 Ιουνίου, συνεπώς από τι 16 Ιουνίου του 2012, απαγορεύεται η αλία για τα ευρωπαϊκά σκάφη στην ΟΣ ε, τη γουινεα Το Συμβούλιο μετά από το πραξικόπημα αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση του πρωτοκόλλου και να αναθεωρήσει από νομική απόψη τα κείμενα ώστε ο φάκελος να είναι έτοιμος από νομικής απόψεως ώστε να μην υπάρχουν αντιρρήσει από τα κράτη-μέλη επί τη ουσία. Ωστόσο, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην λάβει καμία απόφαση μέχρι να επανέλθει η, κατάσταση, η πολιτική κατάσταση στο κανονικό. Εκτότε λοιπόν το έγγραφο βρίσκεται στο Συμβούλιο, γι' αυτό το λόγο δεν έχει το Συμβούλιο ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου επίσημα. Από εκείνη τη στιγμή εμείς έχουμε τακτικές επαφές ε, ως ε, Κομισιόν με την αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί στον Πισάου ώστε να μαθαίνουμε τις πολιτικές εξελίξεις που δυστυχώς προς το παρόν είναι σε αναμονή. Δεν έχουν αναθερμανθεί οι σχέσεις ε, μεταξύ της ε, γωνίας Μπισάου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πράγματα είναι ευαίσθητα και δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε να σε ένα νέο πρωτόκολλο μεταξύ των δύο μερών. Αυτά λοιπόν. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις πιο πρακτικές για την έκθεση της κυρίας ε, ε, αλλά μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον. Απομένει τώρα το Κοινοβούλιο να λαβεί θέση βάσει των ιστορικών του διαδικασιών όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Κύριε Πατράου Νέβες, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω κάποιε παρατηρήσει. Ελέγχθη πρώτα απ' όλα ότι έχουμε αμφιβολίε. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να φτάσουμε τη εργασίε. Όχι, δεν έχουμε αμφιβολίε. Οι αμφιβολίε είναι κάτι το οποίο ασχολούνται η νομική υπηρεσία. Εμεί δεν έχουμε. Επίση, ελέγχθη τι θα κάνουμε. Θα ψηφίσουμε κάτι που δεν θα ε, χρησιμεύει σε τίποτε. Νομίζω δεν είναι λογικό να πει κάτι τέτοιο κάποιο, διότι τα πρωτόκολλα τι περιέχουν. Αυτό που είχαμε πριν, κάποιες μικρές αλλαγές, βλέπουμε τι μπορεί κανείς να αλλιεύσει σε κάθε ζώνη και δεν είναι, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει έτσι τους όρους. Αν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε, ακούστε, ας αποφασίσουμε. Θέλουμε να προχωρήσουμε ή όχι, αλλά όχι βάσει ε, λανθασμένων επιχειρημάτων. Ό,τι κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε θα το κάνουμε βάσει λογικής και επιχειρημάτων. Το λένε αυτό και από την νομική υπηρεσία. Δεν, το να λέμε ότι θα ψηφίσουμε κάτι που δεν θα χρησιμεύσει δεν είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς γίνονται τα πρωτόκολλα, ποια είναι η πραγματικότητα στην Γουινέα Βισάου, ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες αλίας στα ύδατά της, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Λευτικός Στόλος της δεν υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε, όποια και να είναι η πολιτική κατάσταση, βασικά θα είναι όσον αφορά το δικό μας περιεχόμενο το ίδιο. Τώρα, ελέγχθη επίσης ότι δεν είδαμε να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την πολιτική πραγματικότητα. Ειλικρινά πρέπει να πω ότι το γεγονός ότι συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι, ο πρώην και ο τωρινός, στο ε, ΝΟΙΕ, είναι πάρα πολύ θετικό στοιχείο, διότι υπάρχει βούληση, διαλόγου και αλλαγής. Και σε μία τέτοιου είδους κατάσταση, πουθενά δεν συναντώνταν οι πρώην και οι τωρινοί. Και όταν συναντώνταν, σφραγιζόταν με αίμα η συνάντηση. Τώρα λοιπόν που έγινε κάτι τέτοιο, και θέλουν να διαπραγματευτούν μεταξύ τους ότι και δυο θέλουν να αποκατασταθεί η δημοκρατική τάξη του Γουινέα, το βλέπουμε θετικά. Τώρα, υπάρχουν δύο συνάδελφοι εδώ που είπαν μέσα σαφήνεια, όχι, όχι, και κάτι άλλο θέλω να αναφέρω. Αυτός που θα πάρει τα χρήματα ενδεχομένως ε, θα τα χρησιμοποιήσει με στόχο διαφθορά. Ακούστε, από ό,τι ξέρουμε εμείς, παρά τα λίγα στοιχεία που έχουμε, δεν υπάρχει πόλεμος καρτέλ ναρκωτικών, παρά την κατάσταση στην πολιτική. Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα στην οποία ο έλεγχος, η εποπτεία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πιο εύκολους. Γι' αυτό πιστεύω ότι σε σχέση με τη Γουινέα, συγκρινόμενη με άλλες χώρες, έχουμε παράδειγμα χώρες που ξέρουμε πάρα πολύ καλά που πάνε τα χρήματα και ελέγχεται η κατάσταση. Είναι ίσως αυτό κάτι που εκπλήσει κάποιους. Αλλά όντως στη χώρα αυτή βλέπουμε τα χρήματα που αποστέλλονται να χρησιμοποιούνται για να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει. Τώρα, Άκουσα συναδέλφους που λένε καλύτερα σταματήσουμε και μην προχωρήσουμε. Και εδώ θα κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, αυτό το θέμα τέθηκε στις 12 Ιουλίου και μου είπατε κάτι και τώρα μου λέτε κάτι διαφορετικό. Έτσι έχει κατάσταση, δεν έχει αλλάξει. Αν λοιπόν στις 12 Ιουλίου μου είπανε προχώρα, όσο μπορείς να προχωρήσεις, προφανώς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε να πάμε. Και ξέρουμε ότι δεν μπορούσε να υπάρχει επίσημη διαπραγμάτευση. Τώρα, προχωρήσαμε όσο μπορούσαμε. Η Κάρμεν Φράγκα. είναι κρίμα που δεν τόνισε ότι σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε πρόβλημα με την αλληλεία. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε περιμένοντας μία δημοκρατική κυβέρνηση είναι να προχωρήσουμε με λογική μέχρι εκεί που μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά ελέγξαν τον Ιούλιο. Τώρα, ο καθένας πρέπει να πάρουμε τι αποφάσεις, αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ έτσι είχα καταλάβει τα πράγματα τον Ιούλιο και εγώ λέγω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να φτάσουμε, διότι δεν υπάρχει ούτως ή άλλως διαπραγμάτευση με μια δημοκρατική κυβέρνηση και γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Ούτε γιατί μα το επιτρέπει το Συμβούλιο, είτε γιατί δεν μας το επιτρέπει και δεν το λέει η νομική υπηρεσία. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει, η δική μας, που έχουν, που έχει δικός μας αλλιευτικός στόλος. Και πιστεύω ότι επειδή μέχρι τώρα είδαμε ότι χρήματα δόθηκαν, δόθηκαν και σωστά, ε, πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά ανεξάρτητα από αυτά που λέω, θα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση. Ακούστε. Υπάρχει μια διπλή πρόταση. Συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν έχουμε την ικανότητα και αν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Δεδομένου ότι είναι ένα θέμα για το οποίο δεν βιαζόμαστε, να το αφήσουμε να οριμάσει και στην επόμενη συνάντηση οι των πολιτικών ομάδων να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουμε. Ίσως είναι καλύτερα να το αφήσουμε έτσι τα πράγματα. Διότι ε, ούτε θα κερδίσουμε, ούτε θα χάσουμε χρόνο αν το αφήσουμε κατά μέρο προς το παρόν. Και δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Εγώ δεν ξέρω. Τι θέλετε, να το αφήσουμε για να το συζητήσουν στην επόμενη συνάντησή τους οι συντονιστές και η κάθε ομάδα να το δει και με την νομική υπηρεσία, ώστε να έχουμε μια πιο σαφή ιδέα για το αν θέλουμε να συνεχίσουμε, ναι ή όχι. Εντάξει, πολύ καλά. Το επόμενο θέμα μας είναι τα διάφορα, δεν έχουμε τίποτα. Όσον αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών, τις έχετε. Και αν δεν υπάρχει, μπορούμε να τις υιοθετήσουμε. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου, μια ολόκληρη ημέρα. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, σας ευχαριστώ όπως πάντα όλους. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και λύεται η συνεδρίαση.